και θα το ακούσετε και σε ανακοινώσει του Προέδρου, αλλά πρέπει να σας πω τώρα πως υπάρχει πρόβλημα με την δανέζικη διερμηνία. Δεν μπορείτε λοιπόν να ακούσετε δανέζικα. Σας το λέω γιατί όσοι επηρεάζονται από αυτή την έλλειψη θα πρέπει να το έχουν υπόψη τους. Πριν εγκρίνουμε λοιπόν την ημέρα διάταξη, δεν έχουμε διερμηνία από τα δανέζικα. Δεν μπορείτε να ακούσετε δανέζικα, με συγχωρείτε. Έχουμε μία τροποποίηση, το σημείο 7, έγκριση για τον προπολογισμό του 11 θα το αφήσουμε για τον Ιανουάριο. Δηλαδή θα το δούμε στην Επιτροπή στην Επιτροπή όταν αυτή θα συναντηθεί τον Ιανουάριο για την ημερήσια διάταξη. Έχετε κάποιο άλλο θέμα. Όχι, άρα λοιπόν εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Στο σημείο 3 Έχουμε τα πρακτικά, εγκρίνονται. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίρρηση σήμερα, εγκρίνονται και τα πρακτικά. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σας είπα ότι προέκυψε το θέμα αυτό με τα Δανέζικα. Για τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι έχω κάτι να σας ανακοινώσω. Στο σημείο 5, τεχνικά μέτρα και μέτρα ελέγχου στο σκαγεράκι και τροποποίηση του κανονισμού 850 του 98 και του κανονισμού 1342 του 2008. Ξέρετε πως έχουμε μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αντικείμενο συναπόφασης. Ο εισηγητής που την έχει αναλάβει από το ΕΛΚ είναι ο κύριος Κούν και σήμερα θα μας παρουσιάσει το σχέδιο της γνωμοδότησης που μας έχει προετοιμάσει. Έτσι λοιπόν θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Κούν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι για την παρουσίαση αυτό του σχεδίου της Επιτροπής στη διάρκεια της συζήτησης που έγινε. Ε, μετά από αυτή τη συζήτηση πιστεύουμε ότι ορισμένα στοιχεία από πλευράς τεχνικών ε, μέτρων και μέτρων ελέγχου στον πορθμό της Καγεράκης αφορούν την κοινή αλλιευτική πολιτική των μελλοντικών χρόνων. Γι' αυτό το λόγο ε, με τους ε, βοηθούς μου και τους συμβούλους της Επιτροπής ε, σκέφτηκα πώς μπορούν να βρεθούν πρακτικές λύσεις στην περιοχή του Σκαγεράκη. Και αυτές οι πιθανές λύσεις είναι που θα σας παρουσιάσω. Στην τροπολογία 1, στην αιτιολογική σκέψη 1, απλώς και μόνο πρέπει να πούμε, ορίζουμε ποιοι σε αυτή τη ζώνη αλίας ποιοι θα εργαστούν η Δανία, η Σουηδία, η Νορβηγία, τριμερής δηλαδή η συμφωνία μεταξύ των ε, χωρών αυτών, η οποία έληξε τον Αύγουστο έγινε καταγγελία στο 2012 ε, όσον αφορά την πρόταση επιτροπή. και υπάρχει μια ομάδα εργασία που προτείνει μια εναρμόνιση και βελτίωση των τεχνικών μέτρων. Προς το παρόν όμως στη Σκαγεράκη πολλά αλλιεύματα όπως είχε προβλεφθεί μέχρι τώρα απορρίπτονται. Δηλαδή δεν γίνει εκφόρτωση όλων των αλλιευμάτων. Η Νορβηγία έχει υποχρέωση όμως εκφόρτωσης. Η τροπολογία 10, άρθρο 1, 2 και άρθρα 1, 1 2 και 1, 3 αποσαφηνίζεται και συνεπώς ο κανονισμός ισχύει μόνο για τις ζώνες της Καγεράκης που είναι της αρμοδιότητας της Δανίας και της Σουηδίας ως μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ισχύει όμως και για τα σκάφη τα νορβηγικά που αλλιεύουν σε αυτή τη ζώνη. τα κράτη-μέλη ε, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουν ε, ε, δικαιοδοσία στην Νορβηγία οφείλουν να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της Νορβηγίας. Είναι λίγο περίπλοκο το σύστημα, αλλά υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτης χώρας, στην προκειμένη περίπτωση την Νορβηγία. Και συνεπώς η υποχρέωση εκφόρτωση όλων των διευμάτων. Τώρα, στις τροπολογίες 17 έως 20 στο άρθρο 3 και τροπολογία 3 στην αιτιολογική σκέψη 4. Εδώ το, έχω τοποθετηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Πέραν από την υποχρέωση εκφόρτωσης όλων των ε, ειδών της, του 3, προβλέπουν δύο κριτήρια εξαίρεσης. Δηλαδή, ε, τα, οι χθείς στα ψάρια που έχουν ε, μεγάλο ποσοστό επιβίωσης ή όταν ε, το βάρος, το οικονομικό βάρος για τη διαλογή είναι πολύ μεγάλο. Στην τροπολογία 18 περιγράφω σε υπό ποιες προϋποθέσεις η απελευθέρωση ορισμένων ειδών είναι δυνατή. Στην τροπολογία 20 η Επιτροπή θα πρέπει με ορισμένες πράξεις να έχει το δικαίωμα να ορίζει τις προϋποθέσεις απόρριψης ή ελευθέρωσης των ψαριών. Τώρα, όσον αφορά τη διαχείριση των ποσοστώσεων, υπάρχουν οι τροπολογίες 21 και 22 στο άρθρο 4, όπου η Επιτροπή προτείνει όλα τα λιεύματα να καταλογίζονται στις ποσοστώσεις. Αυτή είναι μια καινοτομία στο μέτρο που γνωρίζουμε, όπως ε, κατέδειξαν οι έρευνες, ότι το 20 έως το 30% είχε απορριφθεί στο παρελθόν και κανένα μέτρο εμπιστοσύνη δεν είχε θεσπιστεί σε σχέση με τους αλείς. Το 23 αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο τη πρότασή μου, το οποίο ορίζει ότι αυτή η υποχρέωση εκφόρτωση και ε, απαγόρευση απόρριψη συνδέεται με την αύξηση των ΤΑΚ. Τα κράτη-μέλη όμως θα πρέπει να φροντίσουν ε, να τηρούν αυτή την υποχρέωση. Τώρα η τροπολογία 21 πρόκειται για το κατόφλι ανοχής, δηλαδή πώς ε, ε, θα καθοριστεί σε σχέση με ε, την κατηγορία των ηχθείων και ποια θα είναι τα παρελιεύματα. Εδώ προβλέπουμε 2% ποσοστώσεων που καταλογίζονται, δηλαδή αν θέλουμε να ψαρέψουμε ρέγγα, να υπάρχει ένα ελάχιστο και αν θέλουμε να γίνει διαλογή, αυτό θα κόστιζε πάρα πολύ. Λοιπόν, με 2% μπορούμε να το καταλογίσουμε στι ποσοστώσει. αν είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερη ποσότητα και αν είναι περισσότερα τα είδη, τότε θα έχουμε 5%. Τώρα, για τον γόνο, τα άρθρα 5, τροπολογίες 21 ε, έως 25, η Επιτροπή προτείνει για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εάν δεν υπάρχει ποσοστό επιβίωσης, να χρησιμοποιηθούν μόνο για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Και αυτό όμω είναι μια αντίφαση αφ' αυτού. Τι θα πει για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Δηλαδή, είτε θα τα δώσουμε δωρεάν, είτε πουλείται το ψάρι. Και στη Σκαγεράκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί επειδή οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί οι φιλοκερδείς οργανισμοί, εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν αυτή τη συνήθεια. Τροπολογία άρθρου 6 και η θεολογική σκέψη 7. Η Επιτροπή προτείνει μία απαγόρευση όταν ε, είναι το μάτι ε, μικρότερο των 25 χιλιοστών με εξαίρεση για τα πελαγικά είδη ή τα βιομηχανικά είδη. Εδώ πρέπει να προβλεφθούν 32 χιλιοστά ματιού, επειδή έχουμε όταν υπάρχει το 50% ε, του αλλιεύματος. Αυτή η εξαίρεση ή μάλλον αυτή η προϋπόθεση διευκρινίζεται στην τροπολογία 24. Επειδή όσον αφορά τους κατασκευαστές ειδικών εξοπλισμών ε, αλίες, ήθιστε μέχρι το 90% ενός είδους να το δεχόμαστε, συνεπώς το ποσοστό μας θα πρέπει να είναι μάλλον 80%. Ερχόμαστε ε, σε ένα αποφασιστικό σημείο όσον αφορά τον έλεγχο δηλαδή στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εξ που παίζει αποφασιστικό ρόλο και στην πρόταση της Επιτροπής κυρίως και εδώ έχουμε να κάνουμε τις τροπολογίες 25-31, άρθρο 11, τη σκέψη 12, ορισμένες προκαταρτικές παρατηρήσεις όσον αφορά τον έλεγχο και την εγκατάσταση κάμερας. Εν πλώ, θα πρέπει να καθορίσουμε τις έννοιες με σαφήνεια. Χρειαζόμαστε ορισμούς. Στο άρθρο 2 βλέπουμε REM, Remote Electronic Monitoring, δηλαδή έλεγχος εξ και μιλάμε για τον ανάλογο εξοπλισμό. Κατά τη δική μου άποψη, αυτό το σύστημα REM, δηλαδή ο ηλεκτρονικός έλεγχος εξ γίνεται στο έδαφος και τα κράτη-μέλη θα το αξιολογήσουν και θα το φροντίσουν. Το σύστημα ε, συλλογής και μεταφοράς δεδομένων βρίσκεται πάνω στα σκάφη και διαβιβάζει μόνον τα δεδομένα στο REM και εκτιμώνται, εξολογούνται στο έδαφος. Τώρα, η εγκατάσταση κάμερας στο σκάφος σύμφωνα με το, την έκθεσή μου προβλέπεται ως μη υποχρεωτικό για του ε, τους αλείς. Το κράτος μέλος μπορεί πέραν από την αύξηση των ποσοστώσεων που αναφέρονται για τις, ε, την υποχρέωση εκφόρτωσης, να προβλέψει και άλλα επιπλέον κίνητρα, δηλαδή όταν θέλουμε μια ε, αύξηση, επιπλέον αύξηση των ποσοστώσεων. Αυτό προβλέπεται στο άρθρο 11α. Αυτά τα κίνητρα όμως παρέχονται μόνον στην περίπτωση που τα δεδομένα προβλέπονται και στα ύδατα της Νορβηγίας για παράδειγμα και μεταφέρονται στο σύστημα της παρακολούθησης του ΡΕΜ, δηλαδή, εκτός των νορβηγικών υδάτων. Και υπάρχει υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 3, σε πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, εάν κάποιος ε, παραβαίνει αυτή την υποχρέωση εκφόρτωσης, τότε θα υποχρεωθεί να εγκαταστήσει κάμερες. Εδώ λέμε με σαφήνεια ότι υπάρχει ένα μέτρο εμπιστοσύνης μεταξύ των αρμοδίων αρχών και του επαγγελματικού κλάδου της αλίας. Αρχικά δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά όταν υπάρχουν παραβιάσεις, τότε αυτό γίνεται υποχρέωση όταν, για παράδειγμα, παράβαση, παραβίαση υποχρέωση εκφόρτωση, άρθρο 11α, υπάρχει ένα νέο ορισμό αυτού του συστήματο. Τώρα, για τον μη υποχρεωτικό χαρακτήρα. Το θέμα που τίθεται εδώ σε σχέση με το μήκο των σκαφών, ε, από ποιο μήκο θα πρέπει να βάλουμε ένα σύστημα παρακολούθηση, να εγκαταστήσουμε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, νομίζω ότι το θέμα είναι απλό. Είναι ευνόητο Επίσης, ε, ορισμένα κίνητρα μπορεί να προβλεφθούν ε, για την εγκατάσταση και για τις επενδύσεις. Αυτά πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια. Προς το παρόν έχουμε το 50%, δηλαδή το κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει συγχρηματοδότηση. Η τροπολογία 25. Η μορφή ελέγχων προσδιορίζεται. Είναι ένα πολύ μεγάλο βάρος, επειδή χρειάζεται μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό και γι' αυτό κάνω μια νέα πρόταση, δηλαδή ο έλεγχος να διενεργείται από ένα σύστημα αυτόματης αναγνώρισης. Συνεπώς θα γίνεται αυτόματος έλεγχος. Υπάρχουν ορισμένα συστήματα, σύγχρονα συστήματα αναγνώρισης που μπορούν να αναγνωρίσουν μέχρι ελάχιστο ποσοστό και να επαληθεύουν τα όσα συμβαίνουν. Μπορούμε λοιπόν, αν θέλουμε, να προβλέψουμε ε, την εγκατάσταση ενός συστήματος αυτομάτου ελέγχου που χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά αναγνώρισης. Αυτά παρουσιάζουν κάποιο πλεονέκτημα, διότι ένα τέτοιο σύστημα, όταν εγκατασταθεί στα σκάφη, μπορεί να διαπιστώσει πώς είναι τα αλλιεύματα και δεν χρειάζεται πλέον να γίνεται έλεγχος στην εκφόρτωση και οι ατασθαλίες, οι τυχόν ατασθαλίες μπορούν να επισημανθούν και να παραπεμφθούν στους αλείς οι οποίοι αμέσως μπορούν να παρουσιάσουν αυτά τα στην αγορά με ένα σήμα που να λέει ότι αυτά τα, τα ε, ψάρια έχουν απολυθεί. Την τελευταία φορά είχαμε συζητήσει κατά πόσον υπάρχει αρκετός χρόνος για να αρχίσει ήδη από 1η Πρώτου 2013 να λειτουργεί ένα τέτοιο περίπλοκο σύστημα. Κατά την άποψή μου δεν έχουμε το χρόνο. Επειδή γίνεται η πρώτη συζήτηση έκθεσή μου, ήδη συμβουλεύθηκα τους σχεώδεις συζητητές συζητήσαμε την έκθεση, είδαμε ποιες είναι οι δυνατότητες να υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο έκθεσης, λαμβάνοντα υπόψη ε, τα τεχνικά μέσα που υπάρχουν στο σκαγεράκι. Και πιστεύω ότι αν αρχίσει να ισχύει ο κανονισμό στα μέσα του έτου των ποσοστώσεων, τότε τα πράγματα θα είναι ακόμα πιο περίπλοκα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα αντιμετωπιστούν οι ποσοστώσεις όταν γίνονται εκφορτώσεις ένα κράτος μέλος. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να προβλεφθεί ότι η πρώτη πρώτου του 2014 θα είναι η ημερομηνία της έναρξης ισχύω, διότι πιστεύω ότι ε, οι προθεσμίες είναι πολύ στενές. Ευχαριστώ πολύ τους σκιώδεις συζητητές και ευχαριστώ επίσης τους βοηθούς. Ελπίζω ότι θα βρεθεί μια πολύ καλή λύση για την περιοχή του Σκαγεράκη. Η κυρία Λοβέν παρακαλώ, ευχαριστώ τον ε, κύριο Κούν. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να μιλήσω δανέζικα. Okay. Ε, Θα τα πω στα σουηδικά. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο Κούν για το έργο του, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και έχουμε σημειώσει πρόοδο. Τώρα έχω μια ερώτηση, μάλλον πολλές ερωτήσεις. Τι λέει η Επιτροπή, επιμένει στην πρότασή της ούτω ώστε το 2013 να τεθεί σε ισχύ το κείμενο, γιατί ο κ. Κούν λέει 2014. Τι λέει η Επιτροπή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι καλή ιδέα η δική της. Ας πούμε λέει για 1η Ιουνίου του 2013. Τι πιστεύει η Επιτροπή. Επίσης, σας ερωτώ, πώς μπορούν οι αλληλείς να προπαρασκευαστούν για αυτές τις αλλαγές οι Σουηδοί και οι Δανείοι θα πρέπει να έχουν κάποια εθνική δήμηση για να μπορούν να προσαρμοστούν. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα ούτω ώστε για πρώτη έκτου ή πρώτη εβδόμου να το έχουμε θέσει αυτό σε ισχύ. Αλλά να μου πει και επ' αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιστεύω τώρα κάποια άλλη ερώτηση πάντα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι σημαίνει αυτό το οποίο λέει... Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, το άρθρο... Δεν το βρίσκω, δεν το βρίσκω. Η ιτολογική παράγραφο 4. Άρθρο 3, παράγραφος 4. Εκεί που λέει για κάποιο είδους εξαιρέσεις, παρεκκλήσεις. Λέει για κάποια είδη, προς το ποστό επιβίωσης κλπ. Τι γίνεται όμως με αυτά τα είδη για τα οποία προβλέπει άλλη παρέκκληση, τα οποία δεν προβλέπεται να επιβιώσουν. τι θα κάνουν σχετικά. Οι Ελίες θα πρέπει να ξαναρίξουν τα ψόφια ψάρια στη θάλασσα. Δεν είναι σαφής η ρύθμιση. Προσπάσει ο συνάδελφος Κούν να το διευκρινίσει με την προπολογία του. Αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι σαφής ο σκοπός του εν λόγω άρθρου. Δηλαδή κάποια κάποια ψάρια θα πρέπει να πετάγονται. Τι θα πρέπει να κάνει κανείς με τα είδη τα οποία δεν προβλέπεται να επιβιώσουν. Λέμε τώρα για κάποια κατηξιδότηση πράξη. Ποιος θα αποφασίζει. Οι αλληλείς τι γίνεται για την επιβάρυνση σε σχέση με τα ωφέλη κλπ. Ποιο θα αποφασίσει. Αυτή ήταν η δεύτερη ερώτησή μου. Τώρα, όσον αφορά την πρόταση Κούν. Δηλαδή να δώσουμε επιπλέον ποσοστό σε εκείνους τους αλληλείς, οι οποίοι θα έχουν ε, τέτοιου είδους ε, συσκευές ελέγχου στο σκάφος. αυτές οι πλέον ποσοστώσει από πού θα βρεθούν, μήπως κάποιοι άλλοι θα υποστούν μείωση των ποσοστώσεων. Επίσης, ένα θέμα αρχής, είναι πολύ ε, φιλόσοφες προτάσεις για να προστατεύσουμε επομένως τα ελληνικά αποθέματα, αλλά να δούμε επομένως πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε τις ποσοστώσεις που σήμερα έχουν ε, μοιραστεί στους αλλιείς, Γιατί θα πρέπει να υπάρχει το, η πλέον ποσόστοση. αν θα μείνω στο σημαντικό επίπεδο, τότε ίσως δεν θα πρέπει να είμαι θα υπέρ μιας πιο γρήγορης ε, διανομής πλέον ποσοστώσεων. Ήδη είπαμε ότι έχουμε ξεπεράσει τι ποσοστώσει που μας δίνουν βιωσιμότητα για, το, για τους επομένω. πάρους. Επομένως, ίσως θα πρέπει να βρούμε άλλε, άλλα κίνητρα, άλλα μέτρα για να προωθήσουμε το στόχο μας. Ε, λέμε ότι όλα θα γίνονται για το καλό, τις Αλία, αλλά όμως υπάρχει εδώ πέρα κάποια άλλη αγορά εδώ για, για, για εκείνα τα αλλιεύματα τα οποία θα έπρεπε να, ε, να πραγματοποιούνται. Άρα δεν θα έπρεπε και εμείς να θερμοθετούμε τέτοιες δυνατότητες. Επίσης για το σύστημα τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος επί του σκάφους τι θα γίνει με το κόστος 6 ε, έως 9.000 ευρώ είναι το κόστος λέει για τα σκάφη για να μπορέσουν να καταστήσουν τέτοιες τηλεοράσεις. Άρα πρόκειται εδώ πέρα για πάρα πολλά χρήματα θα πρέπει να επενδύσουν οι αλληλείς. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος επομένως των απορρίψεων. αλλά δεν μπορούσε να υπάρχει κάποιος που να το ελέγχει. Αυτό δεν αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων των αλλιών της ιδιωτικής ζωής. Ε, Πάντω δεν είναι τέτοια ζωή γιατί πρόκειται για χώρο δημόσιο. Πρόκειται για τη θάλασσα που παρακολουθούν οι κάμερε. Και εν πάση περιπτώσει είναι σωστό να ελέγχει κανεί κάποια οικονομική δραστηριότητα σε δημόσιο χώρο. Επομένω, θέλω να συνεννοηθώ για το επόμενο με τον συνάδελφο Κούν. Α πούμε να δούμε τι θα γίνει με τα μεγέθη. Με τα ελάχιστα μεγέθη σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ολιεύματο. Τα είχαμε συζητήσει όταν ε, αρχίσαμε τη συζήτηση για το Σκαλιαράκι. που λοιπόν, θα πρέπει να γίνει κάποιο είδου ε, εναρμόνιση και θα πρέπει να δούμε πώ θα προσεγγίσουμε τι δικέ μα ρυθμίσει με αυτέ τη Νορβηγίας. Και σε αυτό το θέμα του ελαχίστου ε, μεγέθου των ψαριών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μερικοί είπαν ότι πάμε για 40 εκατοστά, είναι στην Νορβηγία 40, αλλά αλλού είναι λιγότερα, Τέλο πάντων είναι 30 στην, ε, στην ε, Δανία, σε Σουηδία και Δανία, Επομένω θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η δυνατότητα αναπαραγωγή των ε, ψαριών. Και για το μερλούκιο και για τα άλλα είδη. Και να γίνει ρύθμιση που να ισχύει και για Νορβηγία και Δανία και Σουηδία. Οπότε ας πούμε οι Σουηδοί ψαράδες λένε ότι θα πρέπει να ανεβάσουμε το όριο. Γιατί τα πιο μεγάλα ψάρια πίθανται σε εμπορία καλύτερα, με καλύτερους όρους. Άρα θα πρέπει μεταξύ Νορβηγίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνει η εναρμόνιση αυτού του ελαχίστου μεγέθους. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κρίστενσεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω πως ε, τελώ υποσύγχυση γιατί είχα σκεφτεί να το πω στα δανέζικα και είναι δύσκολο για μένα να το μεταφράσω έτσι όπως κοιτάω το χαρτί στα αγγλικά. Άκουσα όμως την Ισαβέλα, μίλησε σου ειδικά. Μήπως και εγώ μπορώ να μιλήσω δανέζικα. Γιατί στο κάτω-κάτω παρόμοια γλώσσα είναι. No, if it's possible. Pues si alguien de la interpretación nos lo aclara. Parece que dicen okay. que no. I will make it very brief then. But thank you. Ε, τότε θα είμαι σύντομο αφού δεν Ευχαριστώ πάρα πολύ τον συνάδελφο Κούν για τις προσπάθειες που έκανε σε αυτή την έκθεση και στηρίζω τις περισσότερες από τις τροπολογίες. Αν όμως εξετάσουμε την τροπολογία υπαριθμών 8, δεν μπορώ αυτήν την, ε, το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να το στηρίξω σε θελοντική βάση. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Και για το άρθρο 3 θα ήθελα στο σημείο 5, στο 3, στο 5, στο 14 και στο 20 να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Και αυτό που ζητώ είναι να απαντήσει για το άρθρο 20 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποιο λόγο δίνεται αυτή η ευελιξία για κάθε χρονιά το 20, το 15 και το 10. Δεν θα πρέπει τα ποσοστά να είναι ίδια για όλα τα χρόνια. γιατί η ποσόστοση είναι αυτή κατανέμεται ανά έτος. Αλλά στην ε, ερώτηση αυτή πρέπει να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, ο κ. Ζωπάτση. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν και να σας συγχαρώ, να σας συγχαρώ κύριε Σαγετά γιατί έχετε κάνει πραγματικά άριστη δουλειά. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, λέει ο κύριος Γκρόμπαρτσικ, ε, τις οποίες θα έπρεπε να συζητήσουμε, γιατί νομίζω στα σημεία αυτά θα έπρεπε να μπούμε σε περισσότερο βάθος, ε, τουλάχιστον σχετικά με την έκθεση αυτή. Μέχρι τώρα ε, συζητάμε κάποια τεχνικά μέτρα στο σκαγεράκι. Παρόλα αυτά, αυτά τα οποία δεχόμαστε εδώ, θα επηρεάσουν την Αλία και στη Βαλτική, για παράδειγμα, στην ευρύτερη λοιπόν περιοχή. Άρα λοιπόν η αλλαγή ε, που θα φέρει αυτός ο κανονισμός ε, θα ε, επηρεάσει και άλλα εργαλεία και άλλα αλλιεύματα και άλλες περιοχές. Τεχνικά μου είπατε. Μιλάμε όμως και για βιομηχανική αλία σε κάποιο σημείο. Στη βιομηχανική αλληλεία η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό κλάδο σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης, και όπου ε, πραγματικά επηρεάζει την ζωή των αλλιέων, πρέπει να σας πω πως αυτός ο ελάχιστος οφθαλμός των 32 mm, κατά τη γνώμη μου, των 32 χιλιοστών λοιπόν, θα έπρεπε να συζητηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες. Νομίζω πως θα έπρεπε να εστιάσουμε και σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν την αλληλεία. Δεν ξέρω αν τα 32 αυτά χιλιοστά είναι ο καλύτερος τεχνικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε. Γιατί στην περίπτωση που έχουμε υπεραλίευση κάποιων αποθεμάτων, ενδεχομένως να μην δώσει αποτελέσματα. Ξέρω ότι για την Ρέγκα, για παράδειγμα, σε αυτή την περιοχή, που είναι το είδος που περισσότερο μεταναστεύει μεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και της Βαλτικής Θάλασσας, τα μέτρα αυτά όντως επηρεάζουν την κατάσταση αυτών των αποθεμάτων. Άρα λοιπόν, ας μην μιλάμε μόνο για μέγεθος οφθαλμού, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και κυρίως επαναλαμβάνω όταν αφορά την βιομηχανική αλία. Για τις αποφάσεις που θα πάρουμε, να σας πω πως από αυτές θα εξαρτηθεί το μέλλον της αλίας, όχι μόνο στο Σκαγεράκι, αλλά επαναλαμβάνω και ολόκληρη τη Βαλτική. Κάποια κράτη έχουν ήδη εισάγει τα τελευταία χρόνια ένα σύστημα, ένα σύστημα παρακολούθησης, ένα ηλεκτρονικό tracking. Και πρέπει να σας πω πως έχουμε διαπιστώσει πως δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος της βιομηχανικής αλίας. Τα στοιχεία που έχουμε ε, στη διάθεσή μας δεν είναι αρκετά. Γιατί δεν γνωρίζουμε από ποια περιοχή προέρχονται αυτά τα αποθέματα και επίσης δεν γνωρίζουμε εάν τα στοιχεία αυτά είναι αξιόπιστα τουλάχιστον για τα είδη τα οποία αλλιεύονται στην πραγματικότητα, στην πράξη. Δεν έχουμε λοιπόν καλά στοιχεία γενικότερα για την αλλιεύση που λαμβάνει η χώρα σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω και να ζητήσω και από τον εισηγητή μας να δώσει περισσότερο προσοχή στο θέμα αυτό το οποίο μόλις έθιξα. για τη βιομηχανική αλληλεία και κυρίως για τη ρέγγα. Πρέπει να σας πω ότι στη μεγάλη τους πλειοψηφία μιλάμε για ηχθιάλευρα, ηχθιάλευρα και αυτά τα αλλιεύματα προέρχονται από ύδατα τα οποία είναι εξαιρετική ποιότητα, είναι υγιεινά αλλιεύματα. Θα ήθελα λοιπόν αυτά τα είδη να καταναλώνται και από ανθρώπου. Και νομίζω ότι και αυτό θα έπρεπε να το εισάγουμε στην έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Chairman. Uh, let me start by... Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Κούν για την έκθεσή του και τη σκληρή δουλειά που έγινε σε, μια, σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Ακούσαμε με ενδιαφέρον τις προτινόμενες τροπολογίες και καταλαβα συμφωνούμε ε, με πολλά από αυτά τα θέματα. Τώρα, για ορισμένε τροπολογίες, ίσως θα πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τη σκέψη που βρίσκεται πίσω από τις τροπολογίες. Γι' αυτό θα μας χρειαστούν ορισμένες διευκρινήσεις σχετικά με ορισμένες από τροπολογίες που προτείνονται. Και ελπίζω ότι κατηδίαν διμερός δηλαδή ε, θα δούμε ε, με τον εισηγητή ε, τις απορίες μας ώστε να καταλάβουμε καλύτερα τις τροπολογίες αυτές. Θα ήθελα να αντιδράσω σχετικά με ορισμένα στοιχεία που προκύπτουν από τις προτινόμενες τροπολογίες ή από τη συζήτηση. Ένα από τα θέματα είναι ο χρόνος. Προτείνεται η 1η Πρώτου 2014. Θα ήθελα να σας πω ως Επιτροπή ότι εμείς είχαμε προβλέψει την 1η Πρώτου του 2013 θα άρχισε να ισχύει αλλά θα πρέπει να υπάρχει η συναπόφαση, να εγκριθεί η νέα νομοθεσία ε, με συναπόφαση. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο και γι' αυτό ε, θα πρέπει να το δούμε. Αλλά πιστεύουμε ότι εάν λυθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα στο Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή για να γίνει η υιοθέτηση στη διάρκεια του έτους 2013, τότε η απαγόρευση της απόρριψης μπορεί να αρχίσει να ισχύει από την 1η του 2014. Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσον η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί ώστε να, να υιοθετηθούν τα μέτρα ε, στα μέσα του χρόνου, τον Ιούνιο του 2013 για παράδειγμα. Μπορεί να υπάρξουν όμως ορισμένες δυσκολίες για τους αλληλείς και για τη διοίκηση ώστε να υπάρξει αυτή η απαγόρευση ε, απόρριψης τα μέσα του χρόνου. Θα θέλαμε όμως αυτό το μέτρο να υιοθετηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Μετά από την ε, έγκριση των δύο συνομοθετών αυτή τη πρόταση, τότε θα είμαστε σε θέση να συζητήσουμε την έναρξη ισχύω. Εν πάση περιπτώσει όμω, μπορούμε να δεχθούμε αυτή την, αυτό το χρόνο που επιθυμείτε, 1η Πρώτου 14, για να μην παρακολύεται η διαχείριση ε, της, ε, του αλληλευτικού τομέα στα μέσα του χρόνου. Γενικά, Προτού δούμε τις τροπολογίες, δεν θα σας πω ότι αυτή η πρόταση της, του Σκαγεράκη είναι μια πρόταση που έχει προετοιμαστεί σε περιφερειακό επίπεδο. Γενικά δεν θα έπρεπε να ε, επηρεάσει τη γενική συζήτηση για την απαγόρευση απόρριψης. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η καλύτερη λύση για ε, την απαγόρευση απόρρευση σε αυτό το τομέα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τα μέσα ελέγχου, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα μέσα ελέγχου που έχουν επιλεγεί λαμβάνουν υπόψη τις επιλογές που έχουν κάνει ενδιαφερόμενοι τα κράτη-μέλη ε, της περιοχής ή όταν μιλάμε για το μέγεθος του ματιού ή για το σημείο αναφοράς Όλες αυτές οι έννοιες και όλοι αυτοί οι κανόνες είχαν προταθεί λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα αυτής της περιοχής. Συνεπώς, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για γενικούς κανόνες που θα εφαρμοστούν σε διαφορετικές περιοχές όταν συζητάμε για την γενική απαγόρευση απόρριψης. Ένα άλλο θέμα το οποίο προέκυψε αφορά τα μέσα ελέγχου, τα η χρησιμοποίηση ε, καμερών κλειστού κυκλώματος και καταλαβαίνω πολύ καλά την ανάγκη να σέβεται κανείς ε, τον ιδιωτικό χαρακτήρα και την ιδιωτική ζωή του καθενός, θα πρέπει να, υπάρχει, ε, να υπάρχουν αποτελεσματικές μέθοδοι παρακολούθησης. Η χρησιμοποίηση των συστημάτων κλειστού κυκλώματος είχε επιλεγεί από τα, βασικά, τα δύο βασικά κράτη-μέλη ε, που ενδιαφέρουν για αυτή την περιοχή ως την καλύτερη επιλογή. Η Επιτροπή λοιπόν, και το είδατε στα πλαίσια της μεταρρύθμισης, η Επιτροπή λοιπόν δεν επέβαλε, δεν επιβάλλει την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτού του συστήματος κλειστού κυκλώματος ως γενική υποχρέωση, αλλά προτείνει στα πλαίσια ε, του Σκαγεράκη επειδή ε, αυτό ενδιαφέρει τα, ε, τις περιοχές, ε, τα, τις χώρες εκεί, το, το προτείνουμε ως την καλύτερη επιλογή το σύστημα κάμερας κυκλού κυκλώματος, ε, κλειστού κυκλώματος. Για τη Βαλτική, για παράδειγμα, όταν αυτό το μέσο ελέγχου δεν είχε επιλεγεί από τους ενδιαφερόμενους από τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη ως υποχρεωτικό μέσο τουλάχιστον για τη Βαλτική. Αυτή η υποχρέωση λοιπόν δεν θα είναι γενική, δηλαδή για τον έλεγχο τη απαγόρευση απόρριψη. Αλλά για αυτή την περιοχή, για το πορθμό του Σκαγεράκη, θεωρήθηκε ο καλύτερο τρόπος που θα εξασφαλίζει τον έλεγχο. Η τροπολογία αναφέρεται σε αυτόματο έλεγχο και ηλεκτρονικό έλεγχο. Το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης είναι ένας τρόπος επισήμανσης των ατασταλιών. Είναι ένα από τα μέσα. Δεν υπάρχει αυτοματισμός στον έλεγχο. Και μετά, αφού επισημανθούν τα προβλήματα τότε θα δούμε τι υπάρχει μέσα στην κάμερα, τι έχει καταγράψει η κάμερα. Η κάμερα θεωρείται ως ο καλύτερος τρόπος επισήμανσης των προβλημάτων, των ατασταλιών. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ένας από τους στόχους αυτής της πρότασης είναι να έχουμε τα ίδια μέτρα για όλα τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από τα ύδατα στα οποία πλέουν. Δηλαδή, να μην υπάρχουν άλλοι κανόνες για τα νορβηγικά ύδατα και άλλοι κανόνες για τα ευρωπαϊκά ύδατα. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε να υπάρχουν εναρμονισμένα μέτρα ελέγχου και τεχνικά μέτρα που θα εφαρμόζονται σε όλους που αλλιεύουν στην περιοχή του Σκαγεράκη. Θα πρέπει λοιπόν οι κανόνες να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει τώρα ένα θέμα σχετικά με ε, τις εξαιρέσεις απόρριψης. Θα εξηγήσουμε για ποιο λόγο υπάρχουν οι εξαιρέσεις και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Τώρα θα σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται. πρέπει να καταλάβουμε την τροπολογία που προτείνει ο εισηγητής. Πάλι θα σα εξηγήσω ποια είναι η πρόταση της Επιτροπής. Αναφέραμε ότι υπήρχαν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου ορισμένες απορρίψεις μπορεί να γίνουν δεκτές. Η πρώτη περίπτωση είναι εκείνη όπου υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό επιβίωσης για αυτά τα ψάρια που είναι αντικείμενος απόρριψης. Πρόκειται για ορισμένα είδη, για ορισμένα ψάρια. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. για ψάρια τα οποία μπορούν να επιβιώσουν όταν αλλιεύονται με ορισμένο εξοπλισμό. Μπορεί λοιπόν να προβλεφθεί ε, μία εξαίρεση για αυτά τα ψάρια μόνον όταν αλλιεύονται με ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό αλληλευτικό εξοπλισμό. Θα δούμε λοιπόν τα ποσοστά επιβίωσης και θα πρέπει να γίνει ε, μία εξέταση ε, κάθε είδους ξεχωριστά και στα πλαίσια του κάθε είδους πάλι θα πρέπει να δούμε τι γίνεται ανάλογα με ορισμένους αλληλευτικούς τρόπους. Συμβουλευτήκαμε επιστήμονες για να δούμε ποιες είναι οι περιπτώσεις του υψηλότερου ποσοστού επιβίωσης. Η δεύτερη περίπτωση είναι εκείνη όπου υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες δυσανάλογες. Για παράδειγμα, εκεί όπου υπάρχουν λίγα αντιπροσωπευτικά είδη ε, και όταν υπάρχουν αλλιεύματα αυτών των σπανίων ειδών, εκεί θα μπορούσαμε να μην ζητήσουμε σε έναν αλλιέα να κάνει διαλογή όλων, όλου του αλλιεύματος για να γίνει ξεχωριστή εκφόρτωση αυτών των λίγων ψαριών. Γι' αυτό το λόγο προβλέπεται και εδώ πάλι μια εξαίρεση. Στην τροπολογία δημιουργείται μια σχέση, διασύνδεση με την διατήρηση των ειδών. Εδώ γίνεται λόγος για διατήρηση των ηχθείων, αλλά πιστεύω ότι εδώ πρέπει να καταλάβουμε καλύτερα τι δικαιολογεί αυτή την τροπολογία. Θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους για να εμβαθύνουν τις απαντήσεις σχετικά με τα σημεία κλειδιά που τέθηκαν στη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε ανοιχτοί, είμαστε διατεθειμένες, συνεργαστούμε περισσότερο με τον εισηγητή και θα θέλαμε να έχουμε διευκρινήσεις πάνω σε ορισμένε τοπολογίες, όπως είπα στην αρχή, για να καταλάβουμε πολύ καλά τις τροπολογίες αυτές. Γενικά όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σημαντικό. Μήπως θα μπορούσα να επεκταθώ λίγο για αυτό το οποίο αναφέρθηκε σε σχέση με το άρθρο 3, δηλαδή αυτό το επιπλέον άφθαση στου ψαράδε οι οποίοι θα πρέπει να αποφασίσουν. Κοιτάξτε, το άρθρο 3 συμφωνώ. Δεν είναι πολύ εύστοχα διατυπωμένο γιατί ποτέ δεν θέλαμε αυτό να είναι στην κριτική των αλλιέων και είπαμε ότι αυτό είναι μια ρύθμιση την οποία θα την υιοθετήσει με κάποια κατοξιδότηση πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν θα απόκειται στους αλλήλους να αποφασίσουν σε κάποια συγκεκριμένη έξοδο στη θάλασσα αν θα επιβιώσουν κάποιοι, α, κάποια ψάρια ή όχι. Αν και έτσι φαίνεται από αυτήν την διατύπωση όπως έχει σήμερα το άρθρο 3. Επομένως αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί. Επίσης το άλλο το οποίο έχει δημιουργήσει κάποια σύγχυση είναι αυτό που είπατε για, το, για τις παραπάνω ποσοστώσεις. Εάν κάποιο αλλιεύσει τώρα θα πρέπει να εκφορτώσει όλα αυτά τα οποία προηγουμένω έχει απορρίψει συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ε, άλλων ε, ψαριών τα οποία είναι κάτω από, την από το ε, μέγεθος για να μπορούσαν να διευθυνθούν ομα, αυτέ, αυτές τότε θα πρέπει να αυξηθεί η ποσότητα και δεν πρόκειται για παραπάνω ψάρια δεν θέλουμε να αυξήσουμε το, το, το, το, το συνολικό αλλίευμα. Αυτό που θέλουμε είναι να το μειώσουμε. Και αυτό το οποίο θέλουμε απλώ είναι να προσθέσουμε αυτό το οποίο επρόκειτο να, να, να, να ε, απορριφθεί ε, και αυτό να το βάλουμε στην εκφόρτωση. Άρα θέλουμε ε, να αποφεύγουν τα μικρά ψάρια οι ψαράδες, γιατί δεν επιτρέπεται αυτά να εκφορτωθούν για ανθρώπινη κατανάλωση. Επομένω, έχει αυτό το κίνητρο για να αποφύγει τα μικρά ψάρια. Και επομένω. Ε, τους, αποτρέπουμε από το να ψαρέψουν τα μικρά και στο να ψαρέψουν περισσότερα μεγάλα. Άρα, δεν αυξάνεται λοιπόν. Το, το σύνολο των αλληλευθέντων ψαριών δεν ε, αυξάνεται. Οπότε δεν θέλουμε τίποτα να αυξηθεί η αλλήλευση του, του αλληλευτικού αποθέματος. Θέλουμε να μειωθεί. Αυτό το θέμα βεβαίω μας παραπέμπει και στην άλλη ερώτηση. Τι γίνεται για το, το ελάχιστο μέγεθος των εκφορτωμένων ε, ψαριών. Και αυτό να είναι το, το ελάχιστο μέγεθος ε, για την προστασία των ψαριών. Επομένως, ε, αυτά εδώ τα όρια ίσως δεν είναι αναγκαστικά τα καλύτερα μεγέθη, ίσως τα καλύτερες τιμές θα πρέπει να τις αναθεωρήσουμε, γιατί τώρα μπορεί κανείς αυτά να τα εκφορτώσει, αλλά δεν μπορεί να τα απολύσει. Και επομένως εδώ πέρα έχουμε τα περιθώρια για να δούμε ε, πού θα μπει το κατόφλι. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί μια αγορά για μικρά ψάρια, αλλά την άλλη μεριά δεν θέλουμε και να υπάρχει διασπάθηση κάποιων καθόλου αξιόλογων για κατανάλωση αλληλευμάτων. Άρα θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση αυτού του μεγέθου. Άλλο ερώτημα που υποβλήθηκε για το άρθρο 20 και γιατί έχουμε αυξήσει εδώ την ευελιξία για το πρώτο έτος και κατόπιν πάμε στο 10%. Αυτή η ευελιξία είναι κάτι που μπορεί να είναι χρήσιμο για τους αλληλείς. Γιατί στο τέλος της ε, χρονιάς, αν έχει εξαντλήσει την ποσότητα, μπορεί να πάρει από την επόμενη, μπορεί να μεταφέρει αν έχει και στην επόμενη. Επομένως, μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου μπορεί να γίνει αυτή η κίνηση. Όμω θα πρέπει κανεί να είναι ε, πάρα πολύ προσεκτικό για αυτή την ε, ποσόστοση, γιατί έτσι κανείς προδικάζει κατά κάποιο τρόπο, καταλαμβάνει. Εάν έχουμε μεγάλη ποσόστοση σε μια χρονιά και κατόπιν ε, οι επιστήμονε λένε να γίνει μεγάλη μείωση την επόμενη χρονιά. Εάν επομένω ε, κανεί προδικάσει ότι θα γίνει, ίσω δημιουργήσει δυσκολίε για την κάθε φορά επόμενη χρονιά. Επομένω, είπαμε ότι αυτό το 10% είναι λογικό ποσοστό για κάποιο είδου ε, μακρόπνοη, μακροπρόθεσμη ε, ε, ευελιξία που θα, φορά, θα πηγαίνει από το ένα, μεταφέρουμε από το ένα μέρος, το, από το ένα έτος στο άλλο. Οπότε, είπαμε, περισσότερο ευελιξία από το πρώτο και λιγότερο το δεύτερο έτος, πάμε στο 20%. 15, 10. Αυτό γίνεται γιατί έτσι καθιερώνεται ένα καινούριο καθεστώς για τους αλλιείς οι οποίοι θα πρέπει να εξοικειωθούν στο πώς θα διαχειρίζονται τις ποσοστώσεις που διατίθενται χωρίς να μπορούν να προβούν σε απορρίψεις. Οπότε γι' αυτό και τώρα κάτσαμε και βρήκαμε πώς θα αριστοποιηθούν τα αλλιεύματα σε μεικτό αλλιεύμα με την υποχρέωση της εκφόρτωσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία για να αφομοιωθεί. Επομένως αυτή επομένως ευελιξία είναι για να του δώσει λίγο παραπάνω περιθώριο. Κατά αυτήν την περίοδο, ας το πούμε, εξοικείωση με το σύστημα. Και ε, μετά θα πάμε στο 10% με μακροπρόθεσμα της σχετικής ποσότητας. Και το τέλειο θα ήταν, αν θέλουμε να μετακινηθούμε από το 10%, θα έπρεπε να ρωτήσουμε το Διεθνές ε, Συμβούλιο, το ISIS, ε, να μας πει σε ποιο επίπεδο πρέπει να ορίσουμε αυτή την ενεργειακή τιμή για ούτως ώστε να, έχουμε αποτελεσματικό σύστημα διαχείριση. Δεν θέλουμε να έχουμε υπεραλίωση μακροπρόθεσμα. Επίσης, κάτι άλλο που δεν σας ανέφερα, όσον αφορά την ε, αύξηση στο ΤΑΚ, για να μπορέσουμε να έχουμε την ε, εξισορρόπηση από τις απογρέψεις των απορρίψεων, θα γίνει αυτή η ρύθμιση κατά τα μέσα του 2013 και θα μας πει η ΆΕΣΕΣ τα, τα ΤΑΚ σε ποιο επίπεδο πρέπει να πάνε, ούτως ώστε να παραμείνουμε στο ίδιο επίπεδο εκμετάλλευση του, του, του Και ταυτόχρονα να έχουμε αντισταθμίσει την απαγόρευση των απορρίψεων. Και τα ΤΑΚ δεν θα έχουν σχέση με τα ενήλικα ψάρια, αλλά όπω τώρα, αυτό που μας λέει τώρα η διεθνή οργανισμό, μας λέει ότι το σωμβρό των ψαριών ταξιδίων και 6 ετών. Τώρα, όμω, αυτό το, το, το, το κατώτατο ηλικιακό πρόκειται να μειωθεί και επομένως η Συμβουλή θα αφορά τις καινούργιες ηλικίες. Οπότε θα αυξηθεί το ΤΑΚ. Γιατί συμφωνούν όλοι φαντάζομαι ότι ακόμα και με την απαγόρευση απόρριψης θα υπάρξει ακόμα κάποιο ποσοστό που θα συνεχίσουν να, να απορρίπτουν. Αλλά βέβαια θα έχουμε πολύ λιγότερη, πολύ λιγότερη απόρριψη και άρα θα πρέπει να λειτουργήσουν τα τάκη πέρα των αλλίων. Τώρα, ο στόχος της αύξησης του τάκ είναι να μην είναι τραυματική εμπειρία η απόρριψη των απορρίψεων. Και όταν γίνουμε και με τις προστώσεις αυτές, ε, θα φτάσουμε στα μέσα του έτους και θα έχει πάει πίσω όλη η υπόθεση. Άρα θέλουμε η απαγόρευση αυτή να είναι μια θετική εμπειρία για τους αλληλείς, να είναι κάτι που θα ωφελεί τους πάντες. Συμφωνώ. Η κυρία Λοβέν. Αυτή η αύξηση των ποσοστώσεων δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Δηλαδή, τι θα έχετε, μια συνολική ποσόστοση μια μερική ποσόστοση που θα αυξάνεται. Και η δεύτερη ερώτηση είναι κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε υπόψη τις δοκιμές που έλαβαν χώρα στη Σκωτία, όπου μείωσαν α, στο 0,2% το ποσοστό απορριμμάτων και έτσι βλέπουμε ότι στην περίπτωση που χρειάζεται οι αλληλείς μπορούν να αποφύγουν αυτά τα απορρίμματα, τις απορρίψεις. Θέλετε λοιπόν να αυξήσετε τις, ποσοστε, τις ποσοστώσεις με αυξάνοντας τα ποσοστά για την απόρριψη ή έχετε και μία χαμηλότερη τέτοια ποσόστοση δίνοντας και τη δυνατότητα στους αλληλείς πια να αποφεύγουμε διάφορα μέσα αυτά τα ανεπιθύμητα αλληλεύματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εξετάσαμε με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα διδαχτήκαμε από τις δοκιμές στη Βόρεια Θάλασσα στην ε, Σκοτία, όπου χρησιμοποιούν αυτά τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, που είναι πολύ αποτελεσματικά στην παρακολούθηση των απορρίψεων, των απορριμμάτων. Και εκεί οι αλληλείς πήραν μια επιπλέον ποσόστοση ως κίνητρο για τη συμμετοχή στις δοκιμές. Και βέβαια το ποσοστό αυτή τη ποσότητα ήταν χαμηλότερο από το ποσοστό απόρριψη το οποίο θα γλιτώναμε. Άρα λοιπόν και εδώ μειώνεται η εκμετάλλευση. Άρα περισσότερε εκφορτώσει με ε, μειωμένο ε, τάκ. Αυτό είναι ο στόχο μα. Για τι επιπλέον ποσοστώσει στο Σκαγεράκι θα ζητήσουμε από το Διεθνές Συμβούλιο να μα πει ποια είναι τα ποσοστά αυτή τη στιγμή απορρίψεων και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και πόσο θα μπορούσαμε να προσθέσουμε τα ΤΑΚ χωρίς να αυξήσουμε ε, το συνολικό ποσό απορριμμάτων, ε, απορρίψεων γιατί ε, έχουμε ποσόστοση εκφόρτωση, ουσιαστικά για τέτοιου ποσόστοση ποσόστοση μιλάμε και ό,τι είναι μικρότερο μεγέθους απορρίπτεται. Αυτό που θα προτιμούσαμε εμείς είναι να αυξήσουμε τις εκφορτώσεις αλλά όχι το συνολικά, συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα. Και νομίζω ότι αυτό τους δίνει ένα κίνητρο να αποφεύγουν τα ηχθίδια, γιατί με τον τρόπο αυτό έχουν τη δυνατότητα περισσότερων εκφορτώσεων. Άρα λοιπόν λειτουργεί προς όφελος όλων, αλλά Υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες που θα χρειαστεί να διδαχθούμε ε, από τις δοκιμές αυτές με εξαιρέσεις για κάποια είδη, για παράδειγμα για κάποιους είναι αντιπαραγωγικό για κάποιες εκφορτώσεις, δηλαδή ε, νομίζω ότι μπορεί να αυξήσει κανείς τη θνησιμότητα ε, από κάποιες, ε, σε κάποια είδη αν έχουμε απαγόρευση των απορριμμάτων και να επιβιώνουν καλύτερα αν απλώ δίδεται η δυνατότητα να απορρίπτονται ζωντανά. Ο κύριος Κούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, τους σκιώδες εισηγητές και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω πως τα όσα είπατε και εσείς επιβεβαιώνουν τα δικά μου λεγόμενα και τις τροπολογίες και ε, το ίδιο το κείμενο γιατί αυτή τη στιγμή όταν έχουμε απόρριψη στο 10, 20, 30% ενός τότε τότε χρειάζεται οπωσδήποτε ένα σύστημα το οποίο θα μειώσει αυτά τα ποσοστά. Και θέλουμε βεβαίως και κίνητρα για να αυξηθούν οι εκφορτώσει, ένα κανονισμό για τις εκφορτώσει που θα εφαρμόζεται με τα ποσοστά που μας πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι τέτοιο θα ήταν τέλειο και κάτι αντίστοιχο συνέβη σε αυτές τις δοκιμές στην Σκοτία και αν μπορεί το Συμβούλιο να μας πει ποια είναι τα στατιστικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους για το σκαγεράκι, δηλαδή για το πόσες απορρίψεις γίνονται και τα ποσοστά εκεί, θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε ως σημείο φοιτηρίας. Αν όμως έχουμε κάποιες συνολικές εκφορτώσεις και έχουμε και εκφορτώσεις ειδών που δεν μπορούν να ε, ε, δεν μπορεί κανείς να τα εμπορευτεί, τότε χρειάζεται ένας μηχανισμός έτσι ώστε τα αλλιεύματα αυτά να πηγαίνουν για ηχθιάλευρα για παράδειγμα, να πηγαίνουν σε κάποιες μεταποιητικές μονάδες ή για να ε, χρησιμοποιούνται με κάποιο άλλο τρόπο. Έχουμε μια διμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Η Νορβηγία έχει απαγόρευση εκφορτώσεων εδώ και πολλά χρόνια, αλλά για τα μέτρα ελέγχου δεν επιτρέπει να έχουμε τέτοιου είδους κλειστά κυκλώματα ε, πάνω στα σκάφη. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και εγώ είμαι υπέρ του να είναι εθελοντική η τοποθέτηση αυτών των ε, ε, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα ελέγχεται και το τι γίνεται και θα ελέγχονται και όλες οι ποσοστώσεις. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε συγκεκριμένα αλληλευτικά εργαλεία που θα λαμβάνουν υπόψη τα μεγέθη ε, των ε, ε, ψαριών που επιθυμούμε να εκφορτώνονται. Δηλαδή, για κάποιους τα 30 εκατοστά, για κάποια είδη είναι τάξη. Και εγώ στη Βαλτική έχω ε, ψαρέψει και ξέρω πως κάποια είδη, ε, τα 30 εκατοστά για αυτά είναι εντάξει, η βιομάζα να παράγεται. Και για κάποια είδη νομίζω ότι έχουμε ήδη βρει τις τεχνικές λύσεις. Νομίζω όμως πως η αλληλείς θα πρέπει να είναι η φίλη μας, θα πρέπει να είμαστε σε αυτή την προσπάθεια η συμμαχή μας. Και δεν νομίζω πως χρειάζεται να τα κάνουμε όλα με κατεξουδότηση πράξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσύ ξέρετε ένα κατάλογο ειδών, ότι υπάρχει ένας κατάλογος ειδών με ε, πολύ υψηλό ποσοστό επιβίωσης. Και αυτό που χρειάζεται είναι οι αλληλείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και να αποφασίζουν οι ίδιοι εάν κάποιο είδος έχει υψηλό επίπεδο ε, επιβίωσης ή όχι. Γιατί τι κάνουν πάνω στο σκάφος. Ε, οι ίδιοι διαλέγουν ε, τι θα απορριφθεί. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι και οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι για να είναι βιώσιμη η αλία τους. Τώρα, για τις αρχές αλλά και για τους αλληλείς αυτό που χρειάζεται είναι να εργαστούμε σε μια βάση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Τελείωσε λοιπόν το θέμα αυτό. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Είναι το σημείο 6. Η... Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Μαυρίκιου. Αλληλευτικές δυνατότητες και οικονομική αντιπαροχή. Τώρα για το προηγούμενο σημείο, χρόνος για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 9η του μηνός το μεσημέρι. 9 Ιανουαρίου το μεσημέρι λίγη προθεσμία για τις τροπολογίες. Για το προηγούμενο σημείο και τον Ιανουάριο στην Επιτροπή θα το ψηφίσουμε. Τώρα λοιπόν μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Sí, bueno, confirmar eso que es Στι 9 του μηνό είπα για τι τροπολογίε. σω έλεγε 3 του μηνό, αλλά όχι πλέον για τι τροπολογίε μπορεί να, μπορείτε να τι καταθέσετε μέχρι τι 9 πρώτου. Τώρα για το επόμενο σημείο, το έκτο, που είναι η έκθεση Σάντσε Πρεσέδο. Ο εισηγητή θα μα παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο αυτό, το οποίο μα έχει ε, καταθέσει. Έχετε το λόγο, συνάδελφε. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε πρώτη. Έγινε πρώτη ανταλλαγή απόψεων επομένω όσον αφορά αυτή τη συμφωνία και την ανάλυση του νέου πρωτοκόλλου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία Μαυρικίου. Και είχαμε εξηγήσει ότι υπάρχουν κάποιε αλλιευτικέ και που ξεκίνησαν το 1989 και ε, κατόπιν ε, αυτές ενέπνευσαν το πρωτόκολλο του 2003 έως 2007 ε, όταν έληξε, οπότε όμως δεν έγινε ανανέωση. Και φτάσαμε στις σημερινές διαπραγματεύσεις, οπότε και ε, μόνο γράφει το, το πρωτόκολλο από την Επιτροπή στις 23 Φεβρουαρίου του 2012. Οι νέες προϋποθέσεις που τάσει αυτό το πρωτόκολλο είναι ε, χρηματική αντιπαραχή ψωγραφής είναι 60.000 ευρώ, ε, 5.500 τόνους όπως ούτε αναφορά, το οποίο είναι κάτω από αυτό το οποίο ε, προβλέπεται τώρα. Ε, δηλαδή 6.500. Και έχουμε επίσης 41 την 45 παραδιάρια επιφανείας. Και έτσι είναι εδώ να έχουμε τέτοιου είδους αναθεώρηση σαν δυνατότητα από τα πάνω ή προς τα κάτω. Και επίσης μπορούμε να έχουμε αναθεώρηση και της αντίστοιχης χρηματικής αντιπαραγής. Επομένως οι επιπτώσεις για τον Μαυρίκιο ε, σημαίνουν ότι πρόκειται να ενισχυθεί ο λιευτικός κλάδος ε, αλλά αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι δεν πρόκειται να έχουμε αναγκαστικά αύξηση του συνολικού ε, από, το, από τους Ευρωπαίους στον ε, Ινδικό ωκεανό. θα έχουμε όμως τώρα μια άλλη γεωγραφική κατανομή όσον αφορά τις αλληλευτικές δραστηριότητε και όμως ο Μαυρίκης θα έχει οπωσδήποτε θετική επίδραση γιατί έχουμε 2% της συνολικής εθνικής απασχόλησης και 11.000 θέσεις απασχόλησης που εξαρτώνται από τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε και αυτές οι, ε, συμφωνίες πρόκειται να ενισχύσουν αυτόν τον, ε, τον, ε, τον κλάδο γιατί λέμε και ότι για την αριθμή βιομηχανία που είναι το 15% συνολική των Και έτσι θα τονωθεί η οικονομία τη χώρα. Επίση, έχουμε κάποιε άλλε συγκεκριμένε ρήτρε από το πρωτόκολλο, ρυθμίζει κάποια θέματα όπω την αναθεώρηση ή την αναστολή τη ε, αντιπαραχή. Ε, και είπαμε επίση έχουμε και όρου και προπαθέ και, και ρήτρε σχετικά με ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε έχουμε αυτή την ελευθερική συμφωνία η οποία δεν επηρεάζει πάρα πολύ το σύνολο του προπολογισμού και της οικονομίας του Μαυρικίου. Όμως έχει μεγάλη σημασία όσον αφορά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητα. Όπως είμαστε στη τελευταία μας συνάντηση, στο Μαυρίκιο έχουμε ως αυτό το f 15.000 δολάρια. Και ε, έχουμε περίπου 8% κάτω από το όριο της ένδυας. Έχουμε πάνω σε αυτό το έγγραφο εθνικές στρατηγικές ε, του ε, της ε, Ένωσης και του, του Μαυρικίου για περίοδο 2008-2013 και εκεί προβλέπονται ε, κάποια ωραία πολύ πιο ανεβασμένες σχέση με την, αυτή την συμφωνία, με το ισχύ σύμφωνα και επίσης προβλέπονται, προβλέπονται και κάποιες αλλαγές όταν έχουμε κάποια κατάσταση εκτός της ανάγκης. Επομένως, και η αξιολόγηση, η μελέτη δηλαδή, η σχετική, δηλαδή δεν θα υπάρξει απλώς οικονομικής, περιβαλλοντικής, ε, δυσμενής επίδραση, και οπότε όσον αφορά τα αλλιεύματα του, του μεταναστεύοντος τόνου είπαμε ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση με τα συμφέροντα των τοπικών ε, αλλιών γιατί υπάρχει αυτή η ρήτρα των 15 μιλίων εκεί που ε, επιτρέπεται να αλλιεύουν τα αλλιευτικά σκάφη για να αποθεθούν τα συμφέροντα των τοπικών αλλιών και επομένως η συνολική αξιολόγηση είναι θετική. Επίσης εξηγήσαμε ότι έχουμε λάβει κάποια διευκρίνηση από τους τοπικούς φορείς. Σχετικά με όλο αυτό το, όλη αυτή τη ρύθμιση, πώς θα εφαρμοστεί, όχι τόσο από πλευρά περιεχομένου, αλλά το ότι θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια και περισσότερες ε, διαβουλεύσεις. Και γι' αυτό το λόγο υποβάλει ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμα δεν έχω λάβει την απάντηση, πάντως όμως έτσι κι αλλιώ θεωρώ ότι πρόκειται έτσι να βαθμιστεί η διαφάνεια με τον ε, ανεβασμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον ανεβαθμισμένο του ρόλο. Και οπότε έχουμε αυτή την αξιολόγηση και την θετική σύσταση που λέμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται πλήρω και άμεση για όλα τα στάδια των διαδικασιών. Αυτά πρόεδρε. Ε, όλοι έχουν λάβει αυτό το κείμενο γιατί δεν τα έχουμε συζητήσει. Οπότε δεν προσθέτω τίποτε άλλο, σταματώ εδώ και πρέπει να ακούσω τη γνώμη των υπολείπων συναδέλφων και τη Επιτροπή. Κύριε Περσέδο, ευχαριστούμε. Κυρία Λοβέν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή. Είμαι πολύ ευτυχής που ο εισηγητής διατύπωσε τους ίδιους προβληματισμούς που έχω και εγώ όσον αφορά τους εμπλεκόμενους ε, στο Μαυρίκιο ε, σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης και για την ενημέρωση ε, σχετικά με τη συμφωνία. Και εγώ έχω τις ίδιες ανησυχίες όσον αφορά την κοινωνία των πολιτών, όπως ανέφερε ο συγητής. Εκείνοι που κάνουν ψάρι ενώσεις ψαράδων, ε, όσοι κάνουν ψαροντούφικο κτλ. Βλέπουν λοιπόν και εκείνοι αυτό το πρόβλημα και δεν θέλουμε να επαναληφθούν τα ίδια στο μέλλον. Αυτό όμως έχει να κάνει με την αξιοπιστία και την εικόνα μας. Δηλαδή όταν γίνεται η διαπραγμάτευση αυτών των αλληλευτικών συμφωνιών, όπως λέμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, οι πιο βιώσιμοι κτλ ότι αυτό είναι το ισχυρό μας επιχείρημα για να συνευθυνθούν οι συμφωνίες με τις διάφορες χώρες. Αν μας βλέπουν όμως αρνητικά σε αυτές τις χώρες, τότε αυτό θα είναι αντιπαραγωγικό. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Συνέχεια, σε αυτήν την Επιτροπή, επαναλαμβάνουμε ότι αυτό είναι πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι προσπαθούμε να είμαστε υπερβολικά βιώσιμοι. Και τελικά ε, η ανταγωνιστικότητά μας είναι αρνητική σε σχέση με άλλους αλληλευτικούς τόλους που δεν λαμβάνουν τόσο σοβαρά υπόψη τα θέματα της βιωσιμότητας και της αηφορίας. Εάν θέλουμε λοιπόν να μας δουν πραγματικά βιώσιμους, θα πρέπει ε, να φροντίσουμε ε, ώστε το Κοινοβούλιο η κοινωνία των πολιτών, όλοι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Αυτή λοιπόν η παρατήρηση ήταν πολύ σημαντική. Ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε θίξει πολλές φορές και υπογραμμίζω, στην συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη προβλέπεται ειδική ποσόστοση για τους καρχαρίες. Και αυτό είναι μεγάλο παραλίευμα στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας και είναι περισσότερο παραλίευμα θα έλεγα ε, γίνεται εμπορική εκμετάλλευση από τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Συνεπώς θα πρέπει να το ορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια. Επίσης θα ήθελα πάλι να ρωτήσω την Επιτροπή σχετικά με αυτή την ρήτρα εμπιστευτικότητα που είναι ένα νέο στοιχείο στη νέα γενεά των αλληλευτικών συμφωνιών. Θα ήθελα να μου δοθούν περισσότερες εξηγήσεις, δηλαδή για ποιο λόγο περιλαμβάνονται στις νέες συμφωνίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ολοβέρα. Θέλω να σου βουλευτείς το λόγο. Η την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε τον ε, συγητή για αυτή την ε, έκθεση. Γιατί σχεδόν όλες οι απόψεις που έχουν εκφραστεί θα τις λάβουμε υπόψη. Θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ θετικό στοιχείο. Για όλη αυτή την ε, περιοχή. Ε, επίσης είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και για την ε, περιφερειακή προσέγγιση, την περιφερειακή διάσταση που ότι είναι πολύ σημαντική Και η προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπωσδήποτε και εμείς θα θέλαμε να ε, εξηγήσουμε περισσότερα όσον αφορά τα όσα έχουν ε, εξηγηθεί, όσον αφορά την διαφάνεια, όπως αναφέρατε, οπωσδήποτε και πάντα μπορεί να τα πάμε καλύτερα, αλλά θεωρούμε ότι στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας διαπραγματεύσεων ή ακόμα νωρίτερα, πριν αρχίσουμε τις επαφές με τους Μαυρικιανούς, πάντοτε προσπαθούσαμε να έχουμε την μεγίστη δυνατή διαφάνεια και έτσι προσπαθήσαμε να συμμετάσχουν στη διαβούλευση όλοι όσοι εμπλέκονται. Και στον Μαυρίκη η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επιτέλεσε αξιολογό έργο σχετικά με αυτό και για την αξιολόγηση. Όταν είχαμε την εκ των προτέρων αξιολόγηση, τότε, τότε ε, μπλέξαμε τους τον τοπικό φορέα των ε, αλλιέων, τόσο ώστε να υπάρξουν επαφέ και ανταλλαγέ απόψεων και με εκείνου. Βεβαίω και έχουμε συνοηθεί με το Υπουργείο Αλία του Μαυρικίου αλλά και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα δύο Υπουργεία είχαν τίποτα να κρύψουν. Προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με του εμπλεκομένου όσο ήταν δυνατόν. Στο τέλος δε, όταν μονογράφηκε η συμφωνία, οργανώσαμε αυτή την συνέντευξη τύπου με την υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίση είχαμε και μια τοπική διάσκεψη που είχε οργανωθεί νομίζω τον Μάιο του 2012. Οπότε η περιφερειακή προσέγγιση τότε θίγει και σε σχέση με αυτό επίσης έχουμε ε, εστιάσει την προσοχή μας στα FPA παρά το θέμα του γενικότερο αυτής της διάσκεψης. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με κάθε ευκαιρία ενημερώνουμε, επικοινωνούμε ε, για τα που προς εμπλεκομένους. Αυτά για τη FPA, τη Συμφωνία Σύμπραξης. Τώρα για τους καρχαρίες, για τους καρχαρίες, όπως αναφέρατε, το θέμα αυτό ανεφεί για πρώτη φορά μετά τη μονογραφή τη συμφωνίας, δηλαδή το Μάιο του 2012 με τη Μαδαγασκάρη. Επομένως δεν ήταν δυνατό κατά διαπραγματεύσεις να ληφθεί υπόψη. Πάντως σίγουρα είναι κάτι το οποίο επεξεργαζόμαστε και να δούμε τις επόμενες ε, συμφωνίες πώς αυτό θα ληφθεί υπόψη όπως πρέπει μας με, με τις συμφωνίες με Μοζαμβίκη και Μαδαγασκάρη. Yes, we, we... Απαντήσαμε στους εκλογικούς βουλευτές για την ε, διαφάνεια. Ναι, το κείμενο χτες μου ξεφύγει από την αρμόδια διεύθυνση, αλλά ακόμα ε, ε, επιμένουμε όσον αφορά την αγκαιότητα της διαφάνειας σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες. Για την φορά πάντως να σας τονίσω ότι αυτή η συμφωνία είναι πραγματικά υποφελής για τον Μαυρίκιο στα πλαίσια της περιφέρειας και έτσι να βαθμίζουμε και όχι μόνο τη συνεργασία μας αλλά και την υποστήριξή μας στις χώρες της περιοχής. Γιατί γνωρίζουμε από πλευρά περιφερειακής προαπτικής ότι χρειάζονται τη βοήθεια για να αναπτύξουν τι δυνατότητές τους και να μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ε, ανάγκη της χρηστής διαχείρισης ε, προστατεύσουν τα είδη τους και άρα αλληλένδετο είναι το θέμα αυτό, όχι μόνο με τις άλλες περιφερειακές, τις κοντινές ε, συμφωνίες, αλλά έχει να κάνει και με, με τη διαχείριση και με όλες τις χώρες της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ε, θα δώσω το λόγο και στον εισηγητή για να κλείσει τη συζήτηση. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τις διευκρινήσεις που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα όσα είπε η κυρία Λοβέν και υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είχαμε ήδη θίξει στην προηγούμενη συνάντηση και όπου συμμερίζομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τις απόψεις σας για τους εμπλεκόμενους πρέπει να σας πω πως αυτές οι σχέσεις οι μακροπρόθεσμες είναι μόνο βιώσιμες εάν ισχύουν οι αρχές της διαφάνειας ε, και της διαβούλευσης και νομίζω πως όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν αυτές τις αποφάσεις που λαμβάνονται και να αξιολογούν κατά πόσο οι αποφάσεις αυτές εξυπηρετούν ή όχι τα συμφέροντά τους ε, στον κλάδο και για το λόγο αυτό υποβάλαμε το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε αυτό το χώρο δεν θέλουμε να είμαστε πατερναλιστές, ούτε να σας ελέγξουμε, ούτε να παρεμβαίνουμε. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε σίγουροι πως οι διαδικασίες απόφασης στις οποίες η ε, Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει να ε, ε, υπογράφονται με τα ίδια πρότυπα μέτρα και σταθμά για όλους. Για τους καρχαριές είναι προφανές πω το ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη όπω γίνεται σε άλλε συμφωνίε, θα πρέπει ε, στο κανονιστικό πλαίσιο να εξεταστεί. Γιατί υπάρχει το θέμα των αλλιευμάτων αυτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, στην παρακολούθηση που θα γίνεται, μία online παρακολούθηση όλων των αλλιευμάτων στην περιοχή αυτή. Για την εμπιστευτικότητα, για το απόρριτο που και αυτό είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό θα πρέπει να είναι αποτελεσματικός ο έλεγχος και η συμμόρφωση με τη συμφωνία και παράλληλα θα πρέπει να διατηρήσουμε την δυνατότητα των διαφόρων εταιριών να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπάρχει η εμπιστευτικότητα και το επιχειρηματικό απόρριτο, αλλά χρειάζεται και μια αξιοπιστία. Πρέπει λοιπόν να γίνεται έλεγχος από τις δημόσιες αρχές και στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγουμε να αποκαλύψουμε εμπορικά μυστικά του στόλου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντσες. Να σας πω πως για τις τροπολογίες 3 Ιανουαρίου είναι η καταληκτική προθεσμία. Αφού έληξε και το σημείο αυτό, τελειώσαμε με τη σημερινή ημερήσια διάταξη. Αύριο το πρωί στις 9 ε, δεν είστε πολύ εδώ. Φέρτε αύριο και την κάρτα για τις ψηφοφορίες και μην ξεχνάτε πως πηγαίνουμε στην αίθουσα 5Ε2. Ευχαριστώ πολύ και τα λέμε αύριο το πρωί.